I think we can start. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά στην πρώτη συνεδρίαση αυτή την πρώτη χρονιά και εύχομαι σε όλους σας καλή επιτυχία, ε, σε όλους σας ε, ε, δυναμισμό για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Όσον αφορά τη νέα χρονιά, ευχόμαστε τα καλύτερα. Βεβαίως ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το παρελθόν και εδώ. Ε, θέλω να σας αναφέρω κάτι δυσάρεστο. Ο Φίλιπ Μπρέπον δυστυχώς απεβίωσε κατά τη διάρκεια των γιορτών. Το 99 πρωτοεξελέγει στην άρθρο του Κοινοβουλίου και έκτοτε ήταν μέλος ή αν θέλετε αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής μας, Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και ήδη ε, ήταν ε, μέλος και στην προηγούμενη επιτροπή για τις μεταφορές και τον ε, τουρισμό. Κατά την τελευταία θητή ήταν μεταξύ άλλων εισηγητής για το μέλλον των περιφερειακών αεροδρομίων. Δεν έπαψε να υπογραμμίζει τη σημασία της εδαφικής συνοχής και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στις διάφορες περιοχές συμπεριλαμβανομένων και των West Midlands της γενέτηράς του εκεί όπου γεννήθηκε και τους οποίους εκπροσωπούσε εδώ στο Κοινοβούλιο. Παλαιότερα ήταν εισηγητής για τα ΤΕΝ, τη Μαρκοπόλο, όπως και για το σύστημα των εμπορευματικών μεταφορών. Και επιπλέον ήταν και πολύ ενεργός πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τη σχέση με τον Καναδά. Πρέπει να σας πω, τον Φίλιπ Μπρέπεν τον αντιμετώπιζα πάντα ως ένα ευσυνείδητο ε, εργατικό συνάδελφο, ο οποίος ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την εκλογική του περιφέρεια και εκφράζουμε τα συμμελιπιτήριά μας στην οικογένειά του, στους συγγενείς του και στους φίλους του και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εγερτείτε για ένα λεπτό σιγής. Danke Ihnen. So, wir kommen dann zu dem Tagesordnungspunkt. Περνάμε λοιπόν στο σημείο υπαριθμών 3 τη ημερησία διάταξη. και πρόκειται λοιπόν για την ε, ανακοίνωση του Προεδρίου, της Μεσόλυτα του συμβουλιου πρώτη ανάγνωση σχετικά με την οδηγία για τα βάρη και τις διαστάσει. Και οφείλω να ε, πω και τη θέση του Συμβουλίου. Η θέση Συμβουλίου σχετικά με εκδόση ε, ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του Συμβουλίου 96-53 της 25ης Ιουλίου του 1996 οδηγία για την, τον ορισμό των ανώτατων επιτρεπτών διαστάσεων για οχήματα που μετακινούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε διασυνοριακές μεταφορές. Έτσι λοιπόν η διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης έχει ξεκινήσει επίσημα και ο κύριος Λάιχτ ε, θα καταθέσει την έκθεσή του στις 29 Ιανουαρίου. Θα μπορούσε να το κάνει και σήμερα, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει. Πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 4. Είναι η έγκριση των ε, πρακτικών. Η κυρία Μάισνερ ζήτησε το λόγο. Ο κύριος Λάιχτφριτ ε, μου ανέθεσε να παρουσιάσω εγώ την έκθεση του γιατί ήμουνα ε, πάντα παρούσα στην, στην τριμερή συζήτηση. Όχι, όχι, αργότερα σας δώσω το λόγο στο πλαίσιο της τριμερής συζήτησης. Αν γινόταν να το παρουσιάσετε τώρα, θα σας είχα δώσει το λόγο. Πάμε τώρα στην έγκριση των πρακτικών 1-2 ε, Δεκεμβρίου του 2014. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, θεωρώ ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Και έτσι τώρα πάμε στην ανταλλαγή απόψεων με τον νέο πρόεδρο ε, της, ε, του Οργανισμού Συντηροδρόμων στη συζήτηση με τον κύριο Ντόπλμπαου. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε, που θα συμμετάσχετε στη συζήτησή μας και θα μας παρουσιάσετε σύντομα τους συντηρόδρομους, τα σχέδιά τους. Ε, κύριε Ντόπλμπαου, χαιρόμαστε που ήρθατε και έχετε βέβαια το λόγο. Σας καλωσορίζουμε θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κράμα. για να με κατανοείτε άμεσα περισσότεροι από εσά, θα μιλήσω αγγλικά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής ε, που βρίσκομαι εδώ. Ε, είναι η δέκατη ημέρα ε, όπου έχω αναλάβει το αξίωμά μου, τη θέση μου και πρέπει να σας πω ότι ζούμε μία πολύ ενδιαφέρουσα εποχή γενικότερα για τους σιδηρόδρομους, αλλά και πιο συγκεκριμένα για τον οργανισμό των σιδηροδρόμων. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μου δίνετε η ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Ο τρόπος με τον οποίο έχω ε, δομήσει την ομιλία μου είναι καταρχήν θα αναφερθώ ε, στο άτομό μου, θα μου επιτρέψετε να σας συστηθώ και μετά θα συνεχίσω με το όραμά μου για τους, ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συντηροδρόμων. Ε, θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για ένα σχέδιο και για το επιδιωκόμενο και κατόπιν θα περάσουμε ε, στις συζητήσεις κάποιων σημείων που μας ενδιαφέρουν. Να σας πω λοιπόν το εξής. Είμαι 56 ετών. Είμαι Αυστριακός και σπούδασα φυσική στο Πολυτεχνείο, έχω πτυχίο και διατριβή, διδακτορική διατριβή και ε, εργάστηκα κυρίως ε, στον ιδιωτικό τομέα ε, για πάνω από 25 χρόνια. Είχα πάρα πολλές θέσεις στον τομέα της των προμηθειών και εργάστηκα στην Αυστρία, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σουηδία και τέλος στη Γερμανία. Ανάμεσα σε άλλες θέσεις που κατήχα ήμουν ο επικεφαλής ε, της Bombardier Transport ε, από το 2008 μέχρι το 2013 και πριν από αυτό ήμουν πρόεδρος ε, της, ε, του τμήματος ε, Signaling της Bombardier, σηματοδότηση. Θέλω να σας πω το εξής. Έχω εμπειρία από τη θέση μου που ήμουν πρόεδρος στην Συμβουλευτική Επιτροπή για τους Συνδρομούς στην ΕΡΑΚ. Και σε σχέση βέβαια με αυτό, αλλά περισσότερο σε σχέση με την καινοτομία και με, το, με τη δυνατότητα να αποκτήσω ειδικέ γνώσεις ε, στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήμουν πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής της Shift to Rail από το 2011 έως το 2014. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την πολύ ισχυρή υποστήριξη ε, που προσέφερε η Επιτροπή σας στην πρωτοβουλία Shift Rail. Τώρα, είμαι ευτυχής που είμαι εκτελεστικός διευθυντής τον ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων από την 1η Ιανουαρίου του 2015. Ο Ευρωπαϊκός αυτός οργανισμός είναι ένας σημαντικός οργανισμός ε, που έχει ως στόχο ε, να προάγει το, του σιδηροδρόμου στην Ευρώπη. Το δικό μου το όραμα είναι διτό. Καταρχήν, η αποστολή μας είναι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Και ο δεύτερος στόχος είναι το σύστημα των σιδηροδρόμων να είναι ανταγωνιστικό στον τομέα των μεταφορών. Ανταγωνιστική λοιπόν η σιδηρόδρομη και σε σχέση και με άλλα μέσα μεταφοράς. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ε, ένα εύρυθμα λειτουργούν σύστημα μεταφορών είναι προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και για την ποιότητα ζωής. Επίσης γνωρίζουμε ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι ιδιαίτερα φιλικές προς το περιβάλλον, ενεργειακά αποδοτικές και ασφαλείς. Εκείνο το οποίο πρέπει να ε, μην πάψουμε να επαναλαμβάνουμε είναι ότι πρέπει να γίνει μεταφορά ε, των, του όγκου μεταφορών από άλλα μέσα προς τους ε, σιδηροδρόμους και αυτό θα ήταν μεγάλο όφελος για την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά θα βοηθούσε και στο να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας όπως επίσης και των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα. Ο πρωταρχικός στόχος ε, του, οργανισμού, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων πρωταρχικός στόχος είναι λοιπόν το να συνδράμουν έτσι ώστε να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος ε, χώρος σιδηροδρόμων. Αυτό πάλι σημαίνει ότι τα, οι σειρμοί, οι επιβάτες και τα εμπορέματα να μπορούν να μετακινούνται χωρίς ε, τεχνικούς ή ε, ρυθμιστικούς φραγμούς στην Ευρώπη. Δύο βασικοί στόχοι καθήκοντα των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων είναι η διαλειτουργικότητα, άρα δηλαδή ο οργανισμός είναι αρμόδιος για να καθορίσει τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και δεύτερον είναι αρμόδιος στο να καθορίσει μια κοινή προσέγγιση ως προς την ασφάλεια των κοινών των σιδηροδρόμων. Τέλος, η ε, ευρωπαϊκοί θα καταστήσουν όλο το σύστημα πιο ισχυρό, θα είναι πιο αποτελεσματικοί οι συντηρόδρομοι, θα αρθούν οι τεχνικοί και άλλοι φραγμοί και αυτό πάλι θα οδηγήσει στον περιορισμό ε, του ε, κόστους. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Όταν ε, ο οργανισμός μας, ο ΕΛΑ, θα γίνει μόνο απευθυντική θηρίδα, θα έχει υπάρξει πολύ μεγάλη πρόοδος ή αν θέλετε θα μπορούμε και εμείς να εκδίδουμε πιστοποιητικά για τα οχήματα που θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλοι αυτοί οι στόχοι απαιτούν πολλή δουλειά κατά τα, για τα επόμενα χρόνια και όπως ανάφερα και προηγουμένως ο τεχνικός πυλώνας του πακέτου του τέταρτου πακέτου σιδηροδρόμων ε, είναι καθοριστική σημασία για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Και εδώ λοιπόν και πάλι ε, ζητώ τη βοήθειά σας για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό τον τεχνικό πυλώνα του τέταρτου πακέτου συνδεδρόμων το συντομότερο δυνατόν. Ας δούμε τώρα ποια είναι συγκεκριμένα τα σχέδιά μου. Όταν ξεκίνησα πριν από δύο εβδομάδες στον οργανισμό, είπα στους συνεργάτες μας ότι έχω τρεις βασικούς στόχους. Ο σημαντικότερος είναι εξωστρέφεια. Δηλαδή ο οργανισμός ε, πρέπει να είναι εξωστρεφής, να στρέφει το βλέμμα πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε νέα εξέλιξη και επίσης και να είμαστε ανοιχτοί στο τι παραδείγματο χάρη διαδραματίζεται στην Αποανατολή ή στην Αμερική. Ο δεύτερος ε, στόχος για μένα είναι ότι πρέπει να ε, επιφέρουμε θετικές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα σιδηροδρόμων. Και φτάνω μέσω αυτού στο τρίτο θέμα που θέλω να επιτύχουμε είναι δηλαδή η μέγιστη αποτελεσματικότητα, εσωτερική αποτελεσματικότητα. Όσον αφορά τον πρώτο στόχο ή την πρώτη προτεραιότητα, εργαζόμαστε στο πλαίσιο του τέταρτου πακέτου και στόχος μας είναι να επιτύχουμε ουσιαστική συνεργασία με τους εθνικούς φορείς, τους εθνικούς φορείς ασφάλειας, αλλά και με τους εθνικούς ε, φορείς ε, έρευνας. Ο οργανισμός μας ο ΕΡΑ πρέπει να είναι ο χώρος εκείνος όπου συμπλέουν όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Όσον αφορά στην ασφάλεια, στόχος μου και φιλοδοξία μου είναι να υπάρχει μια ουσιαστική νοοτροπία ασφάλειας ε, και αυτό να επιτευχθεί από κοινού με όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Αυτός, αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της δικαιοσύνης. Δηλαδή δεν πρόκειται για το πώς μπορεί κανείς να τιμωρήσει κάποιους, αλλά πρόκειται για το πώς μπορεί κανείς να αναζητήσει τα αίτια των προβλημάτων και να τα εξαλείψει. Άρα δηλαδή η ασφάλεια, αυτός, αυτή η προσέγγιση πρέπει να βασίζεται στη διαφάνεια, στις έρευνες και επίσης, πόσο μάλλον, στην πρόληψη. Κατόπιν υπάρχει άλλο ένα θέμα που είναι πολύ ενδιαφέρον, το ETTMS, το σύστημα διαχείρισης των σιδηροδρόμων. Και να σας πω ότι ε, παλαιότερα, ήδη από το 92 ασχολούμαι με αυτό το σύστημα, το ERTMS. Αυτό και μόνο δείχνει τις δυσκολίες που υφίστανται, γιατί χρειάστηκαν πάνω από 20 χρόνια έτσι ώστε αυτό το σύστημα το ERTMS να φτάσει στο σύστημα, το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα. Είμαι πεπισμένος ότι δεν ε, μπορούμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Το ERTMS έχει περάσει το μη αναστρέψιμο σημείο και ο δικός μας στόχος είναι να συνεργαστώ με όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη για να επιτύχουμε ένα ε, σταθερό ε, και διαφανές ε, και διαλειτουργικό σύστημα ERTMS. Εμείς, ο οργανισμός μας, είμαστε αρμόδιοι για το σύστημα ERTMS και πρώτο μας καθήκον είναι να καθορίσουμε έναν ε, στρατηγικό χάρτη πορείας για το ERTMS και έχουμε ήδη καθορίσει ένα σημαντικό ε, καθήκον μας είναι να ε, ασχοληθούμε με την ε, ε, baseline 3 του ERTMS. Το επόμενο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαλειτουργικότητα. Και το θέμα το, θα το προσεγγίσω, αν μου επιτρέπετε, ολιστικά. Δηλαδή, όποια αλλαγή στο TSI ή στο καινούργιο TSI θα πρέπει να εξτάζεται κάτω από το πρίσμα της υπεραξίας. δηλαδή αλλαγή συστημάτων μεταφορών θα πρέπει να εξτάζονται κάτω από το πρίσμα της υπεραξίας και των συνεπειών που μπορούν να προκύψουν από οποιοδήποτε κανονισμό. Επίσης, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εργαστούμε για να προχωρήσουμε στο ξεκαθάρισμα των εθνικών κανονισμών. Αυτό για μένα δεν σημαίνει ότι όλα θα τα μεταφέρουμε στα συστήματα μεταφορών, στα TSI. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια όσον αφορά αυτά τα συστήματα. Ε, εκείνο που είναι σημαντικό είναι να ανακαλέσουμε την εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει κατά το παρελθόν. Επίσης, πρέπει να ορίσουμε και τη θέση του Οργανισμού Συνδρόμων ε, στο πλαίσιο ε, της ε, τυποποίησης. Ανέφερα το σύστημα ERTMS. Πρέπει να σας πω ότι η ανάπτυξη αυτού του συστήματος του ERTMS αρχίζει να ισχύει και εκτός Ευρώπης και στην Ασία αν θέλετε. Άρα δηλαδή θα ήταν ε, μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει αρμόδια για αυτό το σύστημα. Όμως ε, πρέπει να ορίσουμε τη θέση μας και στον ε, συντονισμό της έρευνας. Ένα άλλο βασικό θέμα για τον φορέα, πολύ μεγάλη σημασία, έχει σχέση με το να γίνει αποδεκτό το σύστημα των συνδρόμων από την ευρύτερη κοινή γνώμη. Ένα άλλο λοιπόν σημαντικό θέμα είναι ο θόρυβος. Και ε, αυτό πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας. Επίσης, ε, ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνδρόμων έχει διάφορα αρχεία Στόχος μου είναι να τα εξορθολογικεύσω, να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα και αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι να μειωθούν επιπτώσεις ε, για τα κράτη-μέλη. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για το ευρύ κοινό είναι η απλοποίηση της πρόσβασης ε, στους σιδηροδρόμους για τους ε, πελάτες, τους επιβάτες. Και σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του οργανισμού θα προσπαθήσουμε και πάλι να ομογενοποιήσουμε και να απλοποιήσουμε την πρόσβαση αυτή. Θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη επίγνωση των συνεπειών των ενεργειών μας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Σιδηροδρόμων και από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εργαστούμε επί των ορισμών τον καθορισμό δηλαδή της ε, εφαρμογής και παρακολούθησης των ε, βασικών παραγόντων που θα μετρήσουν ιδίω την ε, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας. Και θα πρέπει να εξετάσουμε και την χρησιμότητα του συστήματός μας. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, θα υπάρξει πολύ σοβαρός έλεγχος στις νέες δραστηριότητες τυποποίησης στόχο και σημείο έμφαση σε την διάδοση, την κατάρτιση και διευρυμένη επικοινωνία. Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία του προγράμματος εργασιών μου. Εδώ ίσως θα ήταν καλό να ακούσουμε και τις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. Παρακαλώ, Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στους συναδέλφους ε, για ερωτήσεις. Ο κύριος Βαντερκάμπ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο κ. Δοπελμπάουρ είχε χρόνο να βάλει τα ακουστικά του. Τον καλωσορίζω θερμά. Εντάξει, να σας δώσουμε λίγο χρόνο για τα ακουστικά. Κύριε Ντόπελμπάουερ, ακούτε τώρα τη γερμανική διερμηνία. Ωραία. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας εύχομαι καλή επιτυχία με τη νέα σας θέση και ιδιότητα. Προσωπικά θεωρώ ότι έχουμε υπερβολικά πολλούς νομικούς ε, και τεχνικούς ε, σε αυτούς τους ε, φορείς και είναι καλό το ότι έχουμε και έναν μηχανικό και ειδικό της φυσικής. Ξέρω ότι εργαστήκατε στην Μομπαρδιέ και ότι ξέρετε καλά από τρένα. Καλό είναι λοιπόν τώρα που είστε τώρα και σε όλες τις διαπραγματεύσεις με το, με για το TTIP και την εξαγωγή των τρένων Μομπαρδιέ προς την Αμερική. Ε, σημείωσα όλες σας τις προτεραιότητες, τις οποίες και στηρίζω. Και υπό την ηγεσία του κυρίου Κράμερ ε, με προσμονή βλέπουμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων πριν από το καλοκαίρι. Έχω κάποια ερωτήματα για το ERTMS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της κύκλοφορίες. Κυκλοφορίας. Αν κατάλαβα καλά, θα αναλάβουμε αυτό το ζήτημα το 2016. Είναι ορθό το χρονοδιάγραμμα γιατί βλέπω ότι πολλά επιμέρους κράτη-μέλη δεν έχουν φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο, ιδίως ό,τι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και το επανομαζόμενο request to change. Οι αλλαγές δηλαδή στις τεχνικές προδιαγραφές που συνδέονται με τα εθνικά συστήματα. Θεωρείτε ότι μπορείτε να υλοποιήσετε αυτό το χρονοδιάγραμμα και ποια είναι η αρχική σας εντύπωση μετά από 14 ημέρες. Θα τα καταφέρετε? Αυτά, Πρόεδρε, εν είδη πρώτη παρέμβαση. Ευχαριστώ. Ja, ja, wir teilen uns alles mit dem Kollegen Wim. Ähm, herzlich willkommen, Herr Doppelbauer. Σας καλωσορίζουμε θερμά, κύριε Doppelbau, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία στη δουλειά σας και νομίζω ότι θα συναντιόμαστε συχνά στις Βρυξέλλες. Δείξατε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και νομίζω ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πράγματι να υπάρχει ε, μια σωστή συνεργασία στον τομέα των ε, σιδηροδρόμων και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε ένα κοινό σύστημα σιδηροδρόμων. Ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε λάβει αρκετά μέτρα. Αναφερθήκατε στο τέταρτο πακέτο σιδηροδρόμων, όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, το πλαίσιο των διευρωπαϊκών ε, δικτύων συμφωνήσαμε να υπάρχουν κοινοί διάδρομοι, το συμφωνήσαμε από κοινού με τα κρατημέλη. Και αυτοί οι κοινοί διάδρομοι προβλέπουν και σημαντικά τμήματα ε, με σιδηρόδρομο. Το ERTMS είναι η προϋπόθεση συνεκουανών για να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει βέβαια και το άλλο, ότι ε, στα κράτη-μέλη εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλές αντιρρήσεις στη δική μου την πατρίδα και στο αρμόδιο Υπουργείο γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιοι που διαφορούν παντελώς για το τι αποφασίζουν οι Βρυξέλλες. Οι άνθρωποι δηλαδή παρόλα αυτά εξακολουθούν να κάνουν αυτό που πιστεύουν οι ίδιοι σωστό. Και όσον αφορά το EATMS και στη Γερμανία για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις, ας το πω έτσι προσεκτικά. Βέβαια άλλαξαν εντωμεταξύ τα πράγματα. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Εσείς τι πιστεύετε, θα γίνει κάτι στο Βερολίνο. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που με ενδιαφέρει είναι πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε με το δεύτερο πακέτο σιδηροδρόμων. Το γεγονός ότι είναι πολύ σημαντικό, το έχουμε καταλάβει όλοι, μόνο που ε, και καθαρά πολιτικά υπάρχουν διαφορετικοί στόχοι. Ας το πούμε έξι. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί οι οποίοι αυτό το πολιτικό τμήμα το βρίσκουν ιδιαίτερα σημαντικό. Υπάρχουν όμως και αντιδράσεις, ε, τις ξέρουμε αυτές όλοι μας πάρα πολύ καλά. Στον τεχνικό τομέα είναι το πόλιος. Αυτός ο πολιτικός τομέας ε, αντιμετωπίζεται από κοινού ε, με τον τεχνικό, ο πολιτικός με τον τεχνικό. Πριν από ένα χρόνο είχαμε πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση και αυτό θα πρέπει να το περάσουμε ως κοινό πακέτο. Βεβαίως νομίζω όλοι γνωρίζουν ότι τώρα είμαστε στην τρίτη προεδρία που συζητιέται από το θέμα και δεν έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος. Εγώ εντωμεταξύ πιστεύω ότι το πολιτικό σκέλος, το οποίο βεβαίως και είναι καθοριστική σημασία, αυτό το πολιτικό σκέλος έχει γίνει λιγάκι βάρος, ας το πούμε έτσι. Βάρος που επιβαρύνει εκείνους οι οποίοι επιτιμούν το τεχνικό, ο τεχνικός φάκελος να τελεσφορήσει. Και πολύ σωστά είπατε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε όλα αυτά. Ερωτώ λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές, ο τεχνικός φάκελος πρέπει να αποκοπεί από το πολιτικό σκέλος ε, για να μπορούμε με τον τρόπο αυτό να προχωρήσουμε στο πολιτικό σκέλος. Ε, και αν γίνει αυτό νομίζω ότι ένας χρόνος φτάνει. Έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος ε, Ρόμπερτ Ζήλε. Ε, καλώς ήρθατε κύριε το σε αυτήν την Επιτροπή και συγχαρητήρια με τη, για τη νέα σας ε, θέση ως επικεφαλής του ΕΡΑ. Θα μιλήσω αγγλικά. Είναι δύσκολες οι συγκυρίες για την ΕΡΑ, γιατί τώρα βρισκόμαστε στη φάση ολοκλήρωσης ε, του τεχνικού πυλώνα. Δεν θα θέσω πολιτικά ερωτήματα, γιατί αυτά θα αποφασίσουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτό που μας απασχολεί εμάς είναι η πρόσληψη νέου προσωπικού για τον αέρα, εάν οριστικοποιηθούν όλα αυτά έχετε ολοκληρώσει αυτό το στάδιο, δηλαδή έχετε καθορίσει πόσο άτομα χρειάζεστε και πού θα τα βρείτε αυτά τα άτομα. Δεύτερον, η σχέση σας με, το, με την NSA μετά την έγκριση του τεχνικού πυλώνα, γιατί προφανώς μετά θα υπάρξουν πολλές ε, συμβάσεις με τον NSA και τα κρατη Και υπάρχουν ανησυχίες στα κρατη ότι δεν θα πληρώσετε αρκετά ή ότι θα μεταφέρετε άτομα από τον NSA στον αέρα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις. Υπάρχει πολιτική θέση λοιπόν του επικεφαλής του ΕΡΑ για αυτά τα ζητήματα. Κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Εγώ προέρχομαι από τη Λετωνία. Και πάντα μιλώ για αυτά τα απομονωμένα δίκτυα, όχι μόνο λόγω προεδρίας, γενικά τα αναφέρω. Πριν από ένα χρόνο περίπου υπήρξε μια επίσκεψη και είχαμε ζητήσει αν υπάρχουν πληροφορίες στη βάση δεδομένων σας για τη λειτουργία ε, στη Φιλανδία, Εστονία, Λιθουανία και Φιλανδία. Όχι, λέτε δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτά τα στοιχεία που συνδέονται με το εθνικό πυλώνα. Ποια είναι η επαγγελματική σας γνώμη για την καλύτερη δυνατή λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Δίνεμα, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω θερμά κύριε Ντόπελ Πάουερ, εκ μέρους των φιλελευθέρων στην Επιτροπή Μεταφορών. Έχουν ήδη γίνει πολλά σχόλια, επομένως θα είμαι σύντομη. Είπατε ότι θέλετε έναν ολοκληρωμένο ε, χώρο συνδρομικό στην Ευρώπη και να αυξήσετε και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Και εμεί θα θέλουμε αυτά, θα εργαστούμε λοιπόν από κοινού μαζί σα. Τώρα πιο συγκεκριμένα, είπατε ότι πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία με τι εθνικέ αρχέ. Όμως γνωρίζουμε ότι υπάρχει μία επιφυλακτικότητα, μία αντίσταση και κάποιοι θεωρούν ότι ο αέρα μπορεί να γίνει ένας, ε, μια μορφή υπερδύναμης, υπεροργανισμού. Πώς νομίζετε ότι μπορείτε να κινηθείτε πιο διπλωματικά. Και για το ERTMS είπατε ότι θέλετε να, να το απλοποιήσετε, να απλοποιήσετε την πρόσβαση, αλλά μπορεί να γίνει και οικονομικά προσιτό το ERTMS γιατί ξέρουμε ότι θα κοστίσει ακριβά το ERTMS. Έχετε προτάσεις για το πώς μπορούμε να αποκτήσουμε αυτό το σύστημα πιο γρήγορα, με πιο ομοιόμορφο τρόπο, αλλά και πιο οικονομικά αποδοτικό. γιατί ξέρουμε ότι στη Βαυαρία υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντόπελμπάουερ για την παρουσίασή του. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις νέες σας αρμοδιότητες. Θα ήθελα να θέσω δύο δύσκολα ερωτήματα προς εσάς, υπόψη σας. Ποια είναι η οικονομική κατάσταση του ERA. Έχετε τους πόρους για να διεξακαγεται και να υλοποιήσετε αυτά τα πολύ σημαντικά μέτρα ασφαλείας που έχετε προβλέψει. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας πιο συγκεκριμένα για το τέταρτο συνδεδομικό πακέτο, Ιδίω από την οπτική γωνία της ασφάλειας. Ευχαριστώ. Peter Lundgren. Peter Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε κύριε Ντόπελ Μπάουερ. Άκουσα όσα υπόθηκαν εδώ και συμφωνώ και εγώ με την κριτική που γίνεται στην Ευρώπη. Δεν είναι ο μόνος δρόμος. Μερικές φορές συμβαίνουν περίεργα πράγματα και με τον οργανισμό αυτό σιδηροδρόμων νέρα, ναι, γιατί είναι κάποιοι σε κεντρικό σημείο που αποφασίσουν τι θα γίνει σε εθνικό επίπεδο. Στη Σουηδία, από που προέρχομαι εγώ, έχουμε διάφορα μέτρα και αντιλαμβάνουμε ότι δεν λειτουργούν καλά ε, τα πράγματα από τότε που έχουμε θετήσει τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσον αφορά τη συντήρηση και άλλα προβλήματα θα μπορούσα να αναφέρω την τροφοδότηση σε ηλεκτρισμό, κυρίως το χειμώνα, όπου τα τρένα δεν μπορούν να προχωρήσουν. Δεν μπορούμε δηλαδή να εμπιστευτούμε πια αυτό το σιδηροδρομικό σύστημα. Και έτσι έχουμε την τάση να στρεφόμαστε προς το αυτοκίνητο ή το αεροπλάνο. Εσείς τι λέτε, πώς θα διασφαλίσουμε την καλή λειτουργία των σιδηροδρόμων. Είδατε στην Αγγλία, στη Σουηδία, πώς να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Έχουμε λοιπόν αυτό το συνδρομικό πακέτο τώρα και υπάρχουν διάφορα ζητήματα ανταποκρίσεων, τοπικών μεταφορών που θα χάσουν από αυτό το νέο πακέτο γιατί επικεντρωνόμαστε κυρίως στις κερδοφόρες μεγάλες γραμμές. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα που θα μπορούσα να αναφέρω, τι διαπιστώνω στη χώρα μου. Τι γίνεται με ξένα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν εμπορεύματα. Γιατί πρέπει να δούμε ποια είναι η διαφορά κόστους. Ακόμα υπάρχει μεγάλη διαφορά κόστους. Πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτό το θέμα των ε, μεταφορών εμπορευμάτων από την νότια Σουηδία προς την βόρεια Σουηδία. Γίνεται με φορτηγά και θα στήχιζε πιο φτηνά ίσως αν γινόταν σιδηροδρομικά. Τι θα κάνετε λοιπόν για τον ανταγωνισμό προκειμένου ακριβώς τα τρένε στις δρομικές μεταφορές να είναι ανταγωνιστικές. Ντομινίκ Ρικέ, Κριστίν Βιβονταλόν, Φαντάλεν, Βιλμπάο, Άντερσεν, Μπαχ, Πίπερ, άλλος και κυρία Σμιτ. Και κλείνει ο κατάλογος για να μπορέσει να απαντήσει και ο καλεσμένος μας. Δύο λεπτά καθένας. Ντομινίκ Ρικέ τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε και καλωσορίζω και εγώ τον καλεσμένο μας, τον κύριο Ντόμπλμπάουερ, που έχω εδώ δίπλα μου. Δύο πράγματα θέλω να θίξω γενικά και κάποια πιο συγκεκριμένα για τον οργανισμό. Πέρα από τόσα ανέφεραν οι συνάδελφοι για το τέταρτο συνδρομικό πακέτο. Ποια είναι τα δύο γενικά μου ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν τόσο με τον οργανισμό, αλλά με τη δικιά σας την εμπειρία τι είδους σχέσεις υπολογίζετε να έχετε με τους αντίστοιχους φορείς παγκοσμίω. Κίνα, Ηνωμένε Πολιτείε, Ινδία. Δεύτερον, κατά τη γνώμη σας υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της απόδοσης των σιδηροδρόμων σε σχέση με τις επενδύσεις δηλαδή που κάνουμε. Και ερωτήσεις μου τώρα για τον ίδιο τον οργανισμό. Πρώτο, θεωρείτε ή όχι ότι υπάρχει στρέβλωση ανάμεσα στην αποστολή που δίνει ο νέος κανονισμός στον οργανισμό και το οικονομικό δελτίο που σας έδωσαν. Δηλαδή μήπως σας ζητάνε να μας φέρετε τον ουρανό μετάστρα χωρίς όμως αρκετή χρηματοδότηση. Δεύτερον, πώς βλέπετε εσείς τις σχέσεις με τις εθνικές, ε, τους εθνικούς οργανισμούς ασφάλειας. Νομίζετε ότι η επαφή θα γίνεται με μικρές αντιπροσωπείς ή με μεγάλες. Και τέλος, πιο ειδικά. Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει ένα συμβούλιο ή πολλά συμβούλια για τους διαγωνισμούς μέσα στον οργανισμό αυτόν. Ευχαριστώ. Δεν είχε τελειώσει η μετάφραση στο αυτή μου, λέει ο Πρόεδρο, γι' αυτό δεν σα έδωσα ακόμα το λόγο. Τώρα, κύριε Ρεβό, ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας και ελπίζω και εγώ να έχουμε τακτικές και επικοδομητικές επαφές καθ' όλη τη θητεία μας. Και εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία και ότι καλύτερο για το 2015 που σίγουρα ε, σας επιφυλάσσει πολλή δουλειά. Ξέρουμε την ιστορία, ξέρουμε το τεχνικό σκέλος του τετάρτου πακέτου. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων θέλει να εγγυθεί την ασφάλεια και την διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού χώρου. Όσον αφορά τις πιστοποίησεις τώρα για τις επιχειρήσεις και για τις υποδομές, είναι κάτι πολύτιμο για το μέλλον των σιδηροδρόμων. Οι διαπραγματεύσει γίνονται, όπω ξέρετε, ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο και μένουν ακόμα πολλά να αποσαφινιστούν. Επ' αυτού λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω τα Πρώτον, ποια είναι η άποψή σας για την μεταφορά ε, αρμοδιοτήτων από τις εθνικές υπηρεσίες προς τον αέρα. Το θέμα της μετάβασης, πόσο χρόνο θα κρατήσει, το θέμα της ευθύνη του οργανισμού, των μέσων που διαθέτει ο οργανισμός για να μπορέσει να αναλάβει τις νέες αρμοδιότητες. Κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να κάνουμε ώστε η μεταφορά αυτή να γίνει όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά και διατηρώντας ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Επίσης, πώς βλέπετε εσείς το συντονισμό με τις εθνικές αρχές ασφάλειας προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του ευρωπαϊκού συνδρομικού χώρου και πώς αναλύετε εσείς τις νομικές συνέπειες από τα διάφορα σενάρια μεταφοράς αρμοδιοτήτων, τι επιπτώσεις θα έχουν δηλαδή στις ευθύνε που έχει αναλάβει ο οργανισμός το θέμα της πιστοποίησης και των αδειών σε τι πλαίσιο θα δίνεται, θα δίνεται μόνο από τον ΕΡΑ ή σε κάποιο είδου συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Ευχαριστώ. Πίτερ Φαντάλλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάουερ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Η ομάδα μας είναι πάντα επικριτική απέναντι στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Θέλουμε να δούμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία μιας, ενός τέτοιου οργανισμού. Να αντιληφθούμε τη χρησιμότητά του πέρα από την πολιτική διάσταση. Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις προς εσάς από την εμπειρία που έχετε στο τεχνικό τομέα και γενικότερα στους σιδηροδρόμους. Εγώ ξέρω την Ολλανδία και το Βέλγιο και ξέρω ότι εδώ πέρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε το τρένο το Θύρα, το ξέρετε ίσως, μας ήρθε από την Ιταλία, παραδόθηκε και τελικά είχε πάρα πολλές αδυναμίες ε, το τρένο αυτό. Έγινε πολύ φασαρία και τελικά επεστρέφει και τώρα βρισκόμαστε βέβαια σε νομική διαμάχη. Η ερώτησή μου λοιπόν από αυτού είναι πώς μπορεί να αναμειχθεί στην υπόθεση αυτή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Σκοπεύει να κάνει κάτι για την υπόθεση αυτή. Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε τέτοια περίπτωση άλλη φορά να έχουμε τόσο υψηλών τεχνικών προδιαγραφών τρένο που να μας έρθει με τόσες αδυναμίες. Δεύτερον, όσον αφορά τον ίδιο τον οργανισμό. όσον αφορά το προσωπικό και πού θα εδρεύει. Θα υπάρχουν περισσότεροι χώροι. Πώς θα το διευθετήσετε αυτό. Προκειμένου να συγκεντρωθεί το προσωπικό σε ένα μέρος, αντί να είναι διασπαρμένο. Ευχαριστώ για όλες σας τις εξηγήσεις. Θέλω να ρωτήσω δύο συγκεκριμένα πράγματα εγώ. Ένα από τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποίησαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου οι εθνικές υπηρεσίες να μην έχουν άλλες αρμοδιότητες από αυτές που έχουν τώρα είναι ότι χρειάζονται όλο και περισσότεροι πόροι και προσωπικό για να μπορεί κανείς να αναλάβει την διαθέτηση όλων αυτών των πιστοποίησεων και αδειοδοτήσεων. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτόν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων για να ε, βοηθήσει και να γίνεται πιο αποτελεσματικά το έργο αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω την άποψή σας όσον αφορά τα όσα αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την διαλειτουργικότητα και για τις αρμοδιότητες που θα έχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Πιστεύετε ότι όπως συμβαίνει και με τον Οργανισμό για τις Εναέριες Μεταφορές μπορεί να είναι οικονομικά πιο συμφέρον να έχει περισσότερες αρμοδιότητες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Θα έχουμε δηλαδή το ίδιο αποτέλεσμα όπως έχουμε και με τον Οργανισμό για την και Κυκλοφορία. Έπειτα, είπαμε εδώ στο Κοινοβούλιο ότι τα τέσσερα χρόνια δεν θα φτάνουν σαν μεταβατική περίοδος για να μπορέσει ο οργανισμός ΕΡΑ να έχει μια, ένα κανονικό ρυθμό. Εσείς τι λέτε. Και τι λέτε για το ενιαίο μητρό που θα αποτελεί ένα εργαλείο διαφάνειας. Θέλω να ξέρω ποια είναι η απόψή σας. Τέλος γνωρίζοντας πόσοι δουλεύουν σε κάθε μία από τις εθνικές υπηρεσίες, πιστεύετε ότι για θα ήταν ευκαιρία να αναλάβει όλες τις αρμοδιότητες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις και τις πιστοποίησεις. Ευχαριστώ. Ήθελα να σας συγχαρώ για το έργο της άρα μέχρι τώρα για τις προσπάθειες ε, για επίτευξη περαιτέρω συντονισμού. Ήθελα όμως να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα για τον ε, ρόλο σας ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια, την υπευθυνότητα και τη μυστικότητα. Γιατί είπαμε ότι υπάρχει μια κοινή προσέγγιση ό,τι αφορά την ασφάλεια, αλλά ιδίω στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ανησυχία ότι αν μεταφερθούν σε εσά αυτέ οι αρμοδιότητε σχετικέ με την ασφάλεια, αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο για μα. Ιδίω σε σχέση με τα ζητήματα που άπτονται της ελευθερίας ενημέρωσης για τα ζητήματα ασφάλειας και για κάποια από τα στατιστικά στοιχεία. Δεν ισχύει ότι κάποια στοιχεία που αφορούν ε, απώλειες ε, ζωής ε, δεν καταγράφονται στην Ευρωπαϊκή Βάση ή Είναι κάποια στοιχεία που μας απασχολούν στο Ευρωπαϊκό Βασίλειο. Ξέρω ότι αυτό δεν ισχύει για άλλες χώρες. Και ήθελα να σας ρωτήσω και πιο συγκεκριμένα ε, για το τούνελ της Μάνχης και αν θεωρείτε ότι στο μέλλον θα υπάρχει περαιτέρω ρόλο ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση και ευρωπαϊκή ρύθμιση σε ό,τι αφορά το τούνελ της Μάνχης για την επίλυση κάποιων ζητημάτων ε, που σχετίζονται με τις υποδομές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήλθατε και σας ευχαριστώ και εγώ για τα όσα είπατε. Μιλήσατε για την ασφάλεια, κάτι το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και είναι κάτι που στο οποίο πρέπει να συμμετάσχουν όλοι και δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της πρόληψης. Ε, πολύ σημαντικό. Ωστόσο, με προβληματίζει λίγο η δεύτερη παρατηρήσή σας, γιατί εδώ υπάρχει ένα πολιτικό πλαίσιο που δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα επικοδομητικό εδώ στο Κοινοβούλιο. Πώς να το θέσω διαφορετικά. Δεν είναι όλοι τόσο καλοπροαίρετοι, δεν εύχονται όλοι τα καλύτερα για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Κάποιοι ε, τους βλέπουν ε, ως ε, ένα εμπόδιο, κάτι ιδιαίτερα κοστοβόρο. Εσείς αναλάβετε νέες θερμοδιότητες, όχι μόνο εσείς προσωπικά, αλλά και ο οργανισμός γενικότερα. Πώς θα επιλύσετε αυτό το ζήτημα για να δώσετε μια θετική εντύπωση προς τα έξω για τον οργανισμό. Τι θέση λοιπόν θα λάβει ο ERA σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ κύριο Σπίπερ. Σας έχουμε και εγώ καλή επιτυχία στην νέα θέση. Δύο ερωτήματα. Τα κάτι μελη αρχικά εν μέρει αποδέχονται τις δεξιότητες σας και τα προσόντα σας, αλλά όχι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Δεν ξέρω, το έχετε μελετήσει, τι θα γίνει σε περίπτωση επικέντρωσης αυτών των θέσεων εργασίας. Ποιε θα είναι οι εξοικονομήσεις σε φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, έχουμε εκθέσεις από το 2006 και μετά από το Ελληνικό Συνέδριο που κάθε χρόνο μας λένε γιατί έχει δύο έδρες ο ΕΡΑ. Κάθε χρόνο το Ελληνικό Συνέδριο θέτει αυτή την ε, κριτική. Και υπάρχει αυτό το ζήτημα λοιπόν ε, Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν από πλευράς κόστους πώς μπορούν, μπορεί να γίνεται πιο ε, να εξοικονομήσετε πόρους. Ευχαριστώ κυρία Σμιτ. Ναι, ναι, Βεβαίω, ω Αυστριακή συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες και θέλω να ρωτήσω ε, αυτά που είπε ο συνάδελφος, αυτή η συζήτηση για τις δύο έντρες στο Κοινοβούλιο την έχουμε αυτή τη συζήτηση εδώ και αρκετά χρόνια και από το 2006 ασχολείται και το ελεγκτικό συνέδριο με αυτό. Ερωτώ λοιπόν εσείς θα κάνετε κάτι επ' αυτού. Και το δεύτερο ερώτημά μου απορρέει από αυτά που είπε το ελεγκτικό συνέδριο που είπε ότι όταν προσλαμβάνονται νέοι συνεργάτες δεν υπάρχουν ε, διαφανή κριτήρια και επίση ε, και οι αξιολογήσεις των ε, συναδέλφων και αυτές δεν είναι διαφανής. Εσείς ε, το επιβεβαιώνετε αυτό ή μήπως σκέπτεστε να το αλλάξετε. Πολύ ωραία. Ε, και εγώ ε, τελευταίος ερωτών. Ε, τρία θέματα θέλω να δείξω για τις ε, διαφορετικές έδρες. Ε, βεβαίως και μπορούμε να συζητήσουμε. Δηλαδή ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δύο ε, ε, έδρες. Εγώ έρχομαι από τη Γερμανία και εμείς έχουμε δύο. το 60% είναι στη Βόν και όχι στο Βερολίνο. Γιατί να έχει και ο ΕΡΑ δύο έδρες. να το κάνετε εσείς για να πείστε, πείτε Γερμανούς, να, εμείς τα καταφέραμε μία έδρα, κάντε το και εσείς και να το κάνει και το Κοινοβούλιο. Το δεύτερο που είναι σημαντικό βεβαίως και καθοριστική σημασία είναι ο συμπληρωματικός εξοπλισμός. Ε, άρα δηλαδή, ε, επειδή είναι διασυνοριακές μεταφορές, χρειαζόμαστε ε, ευρωπαϊκή λύση και ο ε, εξοπλισμός, ο συλλογματικός εξοπλισμός είναι καθαριστική σημασία. Είχαμε πει ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια διατίθενται όχι για τον εξοπλισμό αλλά για τις υποδομές. Δέκα δις είχαμε πει στα διευρωπαϊκά δίκτυα και όταν το 80% αλλάζει ε, χρήση χρειαζόμαστε ένα περίπου 80% το θέμα είναι πώς θα μπορέσετε να τα επιτύχετε όλα αυτά. Αναφερθήκατε επίσης στο ERTMS. Εγώ δεν ασχολούμαι τόσο πολύ καιρό όπως εσείς με το σύστημα αυτό, αλλά πριν από 8-9 χρόνια ήμουν εισηγητή για αυτό το σύστημα. Και έγραψα στην έκθεσή μου ότι δεν πρέπει επουδενή με βάση το ERTMS να έχουμε άλλα 20 συμπληρωματικά συστήματα σηματοδότησης. Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουμε 10 χιλιόμετρα ε, αποστάσεις ε, που διανύονται με σύστημα ERTMS. Τα πράγματα όμως δεν έχουν εξυγχρονιστεί. Η καταστροφή είναι η όλη κατάσταση. Ποιος είναι υπεύθυνο για αυτή την καταστροφή και πώς θέλετε να εμποδίσετε να προχωρήσει η κατάσταση. Γιατί το πρόβλημα το γνωρίζουμε εδώ και 10 χρόνια αλλά τίποτα δεν έχει γίνει. Και το τελευταίο. Ο κύριος Ερτούκ ε, έφερε μια νέα λέξη είπε ότι στη Γερμανία υπάρχει ε, διαφορετική προσέγγιση. Καλό το προσέγγιση, όχι προσέγγιση, αντίδραση ήταν, αντίσταση. Οι Γερμανοί, ε, παρότι υπογράφηκε το ΙΡΤΕΜΕΣ, διαφωνούν. Εσείς λοιπόν βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή. Ε, το θέμα είναι το χρειαζόμαστε το σύστημα, γιατί θέλουμε κοινούς σιδηροδρόμους και επενδύουμε, αλλά τελικά όλες οι αρχές σιδηροδρόμων στην Ευρώπη θεωρώ ότι θα επωφεληθούν. Μπορείτε και εσείς να το τεκμηριώσετε με συγκεκριμένους αριθμούς. Ίσως ε, λοιπόν θα ήταν πιο εύκολο να υπάρχουν ε, μόνο δύο σειρμοί ή μορφές τύποι σειρμών στην Ευρώπη και όχι πολλές και πολύ και διαφορετικοί τύποι. Τώρα περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολλές σας ερωτήσεις. Τέσσερις σελίδες έχω σημειώσει εδώ. Κάποιες ερωτήσεις όμως είναι παρόμοιες μεταξύ τους. Και για να πάω από τον κύριο Κράμερ στον κύριο Φαντερκάμπ, θέλω να επανέλθω στο ETRMS. Η ερώτησή σας είχε να κάνει με το σχεδιασμό. Έχω ήδη αρχίσει εντατικέ συζητήσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκα με τον Κάρλ Βίνκ που είναι συντονιστής για το TMS και σήμερα είχα και άλλες επαφές και με την βιομηχανία, με τον κλάδο για να καταλήξω σε συγκεκριμένη άποψη. Εγώ πιστεύω ότι αν μη τι άλλο αυτό που μπορεί να κάνει ο οργανισμός είναι να ειδικεύσει τις, ε, τα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πιστεύω ότι αυτό θα το έχουμε στα μέσα της χρονιάς. Πρότεινε επίσης τον Κάρελ Βίνγκ να καταλήξουμε σε ένα κοινό σχέδιο εφαρμογής γιατί υπάρχουν δραστηριότητες που είναι των οποίων ηγείται ο δικός μου οργανισμός, άλλων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε καλό είναι να έχουμε ένα κοινό πεδίο και άποψη για την κατάσταση για να υπάρχει καλύτερος έλεγχος. προσωπική μου άποψη είναι ότι με τη νέα αυτή πρωτοβουλία και με τη συνεργασία όλων των πλευρών μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου θα πετύχουμε μια ευρωπαϊκή πιστοποίηση, ενιαία. Το οποίο φυσικά μας βοηθάει να εξοικονομήσουμε κόπο και χρήμα. Ενώ όταν έχουμε διαφορετικές εκδοχές, ο κλάδος πρέπει εκ παραλίλου να δουλεύει πάνω σε διαφορετικές προδιαγραφές. Είναι καλό λοιπόν να υπάρχει αναρμόνιση των προδιαγραφών, γιατί τότε θα ελέγχουμε καλύτερα την κατάσταση. Τώρα, έρχομαι πιο συγκεκριμένα στο ζήτημα της Γερμανίας. Πράγματι υπάρχει πολύ θετική συνεργασία από πλευράς της Γερμανίας. Κάτι το οποίο βοηθάει πολύ τις συζητήσεις. Μην το ξεχνάμε, το είπε και η κυρία Μάσεν, ότι είναι από τις χώρες που έχουν μείνει πίσω με το ERTMS, ενώ όλες οι χώρες το εφαρμόζουν. Βέλγιο, Ολλανδία, Αυστρία. Όχι η Γερμανία όμως. Τώρα πιστεύω ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Πώ τώρα στην ερώτηση του κύριου Ερτούκ για το τέταρτο πακέτο. Κατά πόσο θα ήθελα να διαχωριστεί ο πολιτικός πυλώνας από τον τεχνικό θα λέγω ότι δεν είμαι εντελώ ουδέτερος και διάφορος γι' αυτό, γιατί ο τεχνικός πυλώνας και οι νόμοι που βρίσκονται εκεί έχουν να κάνουν με τη δικιά μου δουλειά. Θα ήθελα συνεπώς μια νομική βάση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Υπάρχουν βέβαια καλά επιχειρήματα για να κρατηθούν και οι έξι μαζί. Υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα τον τεχνικό και τον πολιτικό πυλώνα, αλλά η σύνδεση αυτή δεν πιστεύω ότι είναι τόσο ισχυρή ώστε να πρέπει να παραμείνουν μαζί πάση θυσία. Οπότε η απάντησή μου με μια λέξη είναι ναι. Έπειτα υπήρξε μια ερώτηση για το προσωπικό στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνδρομών και τις προσλήψεις. Σύμφωνα με τη σημερινή νομική κατάσταση, ο πρέπει να μειώσει το προσωπικό. 5% μείωση μέχρι το 2050. Αλλά με το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο εμείς πρέπει να αυξήσουμε το προσωπικό. Οργανωνόμαστε λοιπόν. Υπάρχει μια πτυχή που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας έτσι κι αλλιώς. Και έτσι απαντάω και στην ερώτησή σας που λέει πώς θα συνεργαστεί με τις Εθνικές Υπηρεσίες Ασφάλειας ο ΑΕΡΑ και μήπως θέλουμε να φτιάξουμε ένα από πάνω, μια υπηρεσία πάνω από όλες τις άλλες. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να έχουμε δίκτυο, να συνεργαστούμε σε δίκτυο με τις Εθνικές Αρχές Ασφάλειας που θα παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε όλες τις αρμοδιότητες να τις μεταφέρουμε στον αέρα. Πρέπει να είναι δυνατόν οι εθνικές υπηρεσίες ασφάλειας να έχουν κάποια από τα καθήκοντα του αέρα εκείνες. Για μένα υπάρχει εδώ μια πολύ σημαντική πτυχή. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμός Σιδηροδρόμων πρέπει να είναι διατηρητή. Δεν είναι δυνατόν να διαφωνούν δύο εθνικέ υπηρεσίες και να μην μπορούν να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα. Πρέπει να υπάρχει κάποιος που θα ρυθμίζει και που στο τέλος θα παίρνει την απόφαση. Ε, αυτός θα πρέπει να είναι ο Ευρωπαϊκό Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Αλλά όσον αφορά τι αρμοδιότητε. και κοιτώντας την αρχή που διέπει και την ΕΑΖΑ και εκείνος ο οργανισμός συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές. Όσον αφορά το προσωπικό, κάποιοι ευρωβουλευτές εξέφρασαν ανησυχία ότι θα πάρει προσωπικό από τις εθνικές αρχές ασφάλειας ώρα. Πράγματι σκοπεύω να έχουμε μία εκπεριτροπής χρησιμοποίηση του προσωπικού, δηλαδή για ένα κάποιο διάστημα κάποιος από Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας να έρχεται στον αέρα και κάποιος από τον αέρα να πηγαίνει σε μια Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας. Αυτό θα βοηθούσε να λύσουμε το θέμα προσόντων μη αλλά θα λύσει και το θέμα το συναισθηματικό κατά κάποιο τρόπο της συνεργασίας για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε καλύτερα μεταξύ μας. Είχα και μια συγκεκριμένη ερώτηση από αυτή την πλευρά. Ξέρετε ότι προβλέπετε στο τέταρτο συνδρομικό πακέτο να έχουμε συγκεκριμένες συμφωνίες συνεργασίας ανάμεσα τον ΕΡΑ και τις Εθνικές Υπηρεσίες Ασφάλειας εθνικές αρχές ασφάλειας, πιο σωστά. Να ξέρετε ότι εγώ δεν θα αρχίσω με τα πιο περίπλοκα. Ήδη τα συζήτησα αυτά με τον ε, υπεύθυνο της ΥΠΕΘΕΣ ε, και είμαστε σε καλό δρόμο πιστεύω. Θα μάθουμε από αυτή την πρώτη εμπειρία συνεργασίας και έτσι θα προχωρήσουμε. Με ρωτήσατε για ένα ERTMS σε λογικές τιμές. Νομίζω ότι μπορούμε να απλοποιήσουμε, δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε πολλές εκδοχές για διάφορες χώρες. Όταν συνήθως έχει κάνει μεγάλη ποσότητα, ε, είναι και πιο φτηνή. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η εμπειρία που έχω εγώ λέει ότι πρέπει να δίνουμε άδειε σε 12 διαφορετικές χώρες. Αυτές οι 12 διοδοτήσεις για τον ίδιο εξοπλισμό δεν είναι προστιθέμενη αξία. Είναι προστιθέμενο κόστος και προστιθέμενος χρόνος. Αν λοιπόν έχουμε μία μόνο διαδικασία θα είναι πιο φτηνή και θα λειτουργεί αποτελεσματικά. Με ρωτήσατε επίσης για την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Πιστεύω ότι το παράδειγμα αντικατάστασης πολλών και διαφορετικών πιστοποίησεων και αδειών από μία μόνο ε, φτάνει σαν ε, αιτιολόγηση. Όντως είναι προστιθέμενη αξία λοιπόν αέρα. Πρέπει να έρθω τώρα και στο ζήτημα των ε, δύο εδρών, των δύο χώρων εργασίας. Αναρωτήθηκα κι εγώ όταν ε, έφτασα στον αέρα. Αλλά μου είπαν επίσης ότι εγώ που θα είμαι εκτελεστικός διευθυντής δεν θα έχω καμία εξουσία από αυτού. Είναι απόφαση των χωρών μελών. Οπότε πιστεύω ότι το πολιτικό επίπεδο είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει. Εμείς θα ακολουθήσουμε. Πρέπει επίσης να πω ότι δύο χώροι εργασίας, βασικά είναι ένας όπου έχουμε τα γραφεία μας και άλλος είναι στη Λίλ. Είναι δηλαδή ο χώρος στον οποίο πηγαίνουμε και συναντάμε τους συμμετόχους μας, όπου δηλαδή συνεδριάζουμε πιο πολύ. Αν αποφασίσει ο αέρα ότι θα είναι Λίλ Βαλανσιέν, έχει καλώ. Αν είναι κάτι άλλο, ευχαρίστω να το συζητήσω. Θα είμαι στην διάθεσή σα. Ας έρθω τώρα στην ερώτηση τη κύρια Άντερσον για την ασφάλεια και την σχετική προσέγγιση του Ηνωμένο Βασίλειο. Πρώτα απ' όλα, όπως είπα και πριν, θα κάνουμε τα πάντα σε συνεργασία με τα διαφερόμενα μέρη, με τους συμμετέχοντες δηλαδή, θα φροντίσουμε να μην υπάρξει καθόλου απώλεια σε σχέση με τις πληροφορίες που θέλετε στον Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Πάντως, ακριβώς επειδή υπάρχει νοτροπία αυτή ασφάλειας, εμείς τρεφόμαστε προς το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κάνει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια και θέλουμε να αποφεληθούμε και εμείς από αυτήν. Η οικονομική κατάσταση τώρα του οργανισμού είναι κάτι το οποίο έφυξα. Ακόμα περιοριζόμαστε από την προηγούμενη νομική κατάσταση, η οποία μας υποχρεώνει να περιορίζουμε το προσωπικό, να το μειώνουμε μάλιστα, αλλά εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε για το τέταρτο συνεργονομικό πακέτο. Οπότε, περιμένω ότι θα αλλάξει η κατάσταση πολύ σύντομα. Και από τη Σουηδία, αν δεν απατώμε, με ρωτήσατε για τις συνέπειες του τέταρτου σιδηροδρομικού πακέτου. Πρώτα απ' όλα είπατε ότι σας ανησυχεί το θέμα του ανταγωνισμού από τις οδικές μεταφορές, τη μεταφορά εμπορευμάτων δηλαδή οδικός. Μας στόχος του ΕΡΑ είναι ακριβώς οι σιδηρόδρομοι να είναι πιο ανταγωνιστική. Πρέπει να κάνουμε δηλαδή ό,τι μπορούμε προκειμένου η μεταφορά σιδηροδρομικός να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τα φορτηγά και τα εμπορεύματα να συμφέρει να μεταφέρονται σιδηροδρομικός από ό,τι με φορτηγά. Έχουμε έναν σιδηροδρομικό χώρο χωρίς σύνορα, άρα πρέπει να είμαστε σε θέση να μειώσουμε το κόστος και την αδειοδότηση και την πιστοποίηση να τα κάνουμε πιο φθηνά για να έχουμε και οικονομία και καλύτερη ανταγωνιστικότητα. Αναφερθήκατε και στους δεδεμένους σιδηροδρόμους. Κατά τη γνώμη μου, μπορούμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί οι σιδηρόδρομοι από ότι οδικές μεταφορές και μπορούμε να γίνουμε και πιο ελκυστικοί. Έρχομαι τώρα στην θέση μας παγκοσμίω. Όπως είπα, θέλουμε τις επαφές ήδη με το FRA και με την Κίνα θέλουμε να έχουμε επαφές για να καθορίσουμε τη θέση μας στον κόσμο αναφέρθηκα οι και στις σχέσεις μας με τις εθνικές αρχές ασφάλειας. Είναι στο μυαλό μας η συνεργασία και αμοιβή εμπιστοσύνη. Μεταφορά αρμοδιοτήτων, όπως είπα και πριν, μεταφορά αποσπάσεις δηλαδή από τις εθνικές αρχές στον αέρα και από τον αέρα στις εθνικές αρχές ασφάλειας. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο με τον ΕΡΑ που θα είναι ο ενίος φορέας αδειοδοτήσεων και πιστοποίησεων θα αλλάξει την κατάσταση και πρέπει να είναι όλοι προετοιμασμένοι. Και κυρίως ο ίδιος αέρα. Ο κύριος Κράμερ βλέπω ότι κοιτάει το ρολόι του. Οπότε πρέπει να ολοκληρώσω κι εγώ πώς μπορούμε να μεταφέρουμε τα θετικά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Πώς μπορούμε να κάνουμε γνωστό τον οργανισμό αυτό ως έναν αποτελεσματικό οργανισμό. Εδώ είναι θέμα προβολής, είναι θέμα επικοινωνίας και συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Θα φροντίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε τέτοια συγκεκριμένα αποτελέσματα και όταν θα έχουμε κάτι θετικό θα φροντίζουμε να το κοινωνούμε και στο κοινό, να το μεταφέρουμε, να το μαθαίνει ο κόσμος, να το προβάλλουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Έχουμε μια πολύ καλή ιστοσελίδα και θα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα μέσα για να προβάλλουμε ακόμα περισσότερο το έργο του οργανισμού. Ελπίζω να κάλυψα το 80% τουλάχιστον των ερωτήσεων σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ντόπελπαου. Προφανώς και εμείς προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία. Αυτό ήταν το πρώτο και καλό βήμα και είμαι αισιόδοξο ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Πριν λοιπόν κλείσουμε αυτή την ε, ανοιχτή συζήτηση θα ήθελα να χαιρετήσω θερμά ε, τους βουλευτές από τη Γερμανία, από την ε, Επιτροπή Μεταφορών. Κάθονται πίσω-πίσω. Ήταν βέβαια ε, στο τέλος και δεν μπόρεσαν να ακούσουν αυτά που ελέγχθησαν και τη Γερμανία. Κρίμα. Ο κύριος Αρτούκ που σας κάλεσε θα σας τα πει. Σας καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν έρχονται τα Εθνικά Κοινοβούλια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντίστροφα βέβαια. Καλωσορίσατε. και λυπάμαι πάρα πολύ. Ε, τώρα πρέπει να κλείσουμε την ανοιχτή, τη δημόσια συζήτηση, γιατί έχουμε μία συζήτηση για τις ε, τριμερείς ε, συναντήσεις και αυτή γίνεται και κλεισμένη των θυρών, ε, στην οποία συμμετέχουν μόνο ευρωβουλευτές. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά τι να κάνουμε, έτσι το είχαμε προβλέψει για σήμερα. Ευχαριστώ.